να δημιουργήσουμε και εταιρικέ σχέσεις μεταξύ Ιδρυμάτων. Σας ευχαριστώ κύριε Τόκερ και πάλι για την θετική προσέγγισή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κυρίες και κύριοι, εδώ τελείωσε η συζήτησή μας και η ψηφοφορία προβλέπεται για αύριο στις 12. Το τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης είναι η έκθεση της κυρίας Τικάου για μια ανταγωνιστική ψηφιακή ενιαία αγορά η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ως αιχμή του δόρατος. Το λόγο έχει η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το 2010 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οθέτει στρατηγική 2020 η οποία έχει στόχο στην αηφόρο ανάπτυξη και στη βελτίωση της οικονομικής ε, της διακυβέρνησης. Μία από τις βασικές πρωτοβουλίες αυτής της στρατηγικής είναι μια ψηφιακή ατζέντα για την Ευρώπη, μια στρατηγική για τη διερεύνηση του δυναμικού ε, που απορρέει από την εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών. Το Κοινοβούλιο χαιρετίζει την υιοθέτηση του προγράμματος αυτού του στα πλαίσια της στρατηγικής διαλειτουργικότητας και του πλαισίου διαλειτουργικότητας για τι ευρωπαϊκέ δημόσιες υπηρεσίες και ζητάει από τις χώρες μέρη να ευθυγραμμίσουν τις εθνικές στρατιστικέ με τι ευρωπαϊκές πολιτικές. Οι υπηρεσίες αυτές είναι σημαντικές για τη μείωση του κόστους για τη διακρατική διαλειτουργικότητα και για τη δημιουργία της ενιαίας αγοράς. Από επειδή η αγορά κρατικών προμηθειών ε, ε, ε, είναι το 60% και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι το 90% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην διακρατική διαλειτουργικότητα από την άποψη των ε, ε, κρατικών προμηθειών και των ηλεκτρονικών συστημάτων. Αυτό το σύστημα θα υπάρχει παντού και θα χρησιμοποιηθεί καλύτερα. Και αυτό θα συμβάλλει σε μια μείωση κατά 30% του κόστου των κρατικών προμηθειών. Ε, Παρόλο που ε, συμβαίνει αυτό, 14 και 15 χώρες βρίσκονται στην αρχική φάση δημιουργίας αυτών των προγραμμάτων. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία της Ζαμία, της Φιλανδίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας να κάνουν υποχρεωτική την ηλεκτρονική τιμολόγηση και ζητάω η τιμολόγηση αυτή να γίνει υποχρεωτική για όλες τις κρατικές προμήθειες μέχρι το 2016. Βασικά θέματα όπως η διαχείριση ηλεκτρονικής ταυτότητας, η διελικότητα και τα νικητά πρότυπα αποτελούν προϋποθέσεις για μια επιτυχή ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τη διαλειτουργικότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι χώρες μέλη θα πρέπει να επανεξετάσουν τα προαπαιτούμενα σε ό,τι αφορά την ηλεκτρονική υπογραφή για να μπορέσουν να εξαλείψουν όλα τα εμπόδια για τις διακρατικές υπηρεσίες. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το συντομότερο δυνατόν την οδηγία για την ηλεκτρονική υπογραφή για να αυξηθεί η διακρατική διαλειτουργική των ηλεκτρονικών συστημάτων απόδειξης γνησιότητας καθώς και την απόφαση που προβλέπει την αμοιβαία αναγνώριση της Ευρωπαϊκής Απόδειξης Γνησιότητας και Ευρωπαϊκής Υπογραφής. Τα, κοινοβούλια τονίζουν ότι οι διακρατικές διακτηρικές υπηρεσίες θα πρέπει να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν ένα λειτουργικό ε, πλαίσιο για, ε, σε μια αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στι υπηρεσίε. Θα πρέπει να εξυγχρονίσουμε τι υποδομέ ε, τη ηλεκτρονική διακυβέρνηση ε, και τι υπηρεσίε online. Μια ασφαλής, ένα ασφαλές διακρατικό σύστημα αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την προστασία των σημαντικών υποδομών. Χαιρετίζουμε τη συμβολή προγραμμάτων όπως IDA, IDABC, καθώς και την πρακτική πρακτική τους μορφή για τη δημιουργία του, της ε, διαλειτουργικών λύσεων. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει την πρόταση που έχει τίτλο «Συνδέοντας την Ευρώπη», η οποία παρέχει 9 δισεκατομμύρια ευρώ για δίκτυα ευρεία κλίμακας και για ευρωπαϊκές υπηρεσίες δικτύων. Οι μηχανισμοί διασύνδεση θα παράσχουν τη χρηματοδότηση για να μπορέσουν να δημιουργηθούν οι υποδομέ που θα επιτρέψουν τι ηλεκτρονικέ υπηρεσίε απόδειξη γνησιότητα, ε, ηλεκτρονική δικαιοσύνη, ηλεκτρονική υγεία, ηλεκτρονικέ τελωνικέ υπηρεσίε και αυτέ οι υποδομέ θα πρέπει να συμβάλλουν στην διαλειτουργικότητα και να καλύψουν το κόστο συμμετάλληλη σε ευρωπαϊκό επίπεδο διασυνδέοντα υποδομέ των χωρών μελών. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ για την εισαγωγή. Ξεκινάει το Catch the Eye. Έχω 7 ομιλητές. Πρώτος ομιλητής, ο κύριος Παπα-Νικολάου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Ε, θα πρέπει να κάνουμε στο θέμα αυτό μια γενική παραδοχή, η οποία είναι ιδιαίτερος κρίσιμη και η οποία θα κατευθύνει και τις μελλοντικέ πολιτικές μας στον τομέα αυτό σήμερα μέσα σε ένα πολύ βαρύ οικονομικό περιβάλλον διαπιστώνονται μεταξύ των κρατών μελών αποκλίσεις όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών από το διαδίκτυο και με τη σειρά τους αυτές οι διαφορές δημιουργούν σημαντικό χάσμα ανταγωνιστικότητας. δεν είναι λοιπόν μόνο το εργατικό κόστος δεν είναι μόνο οι γενικές δημοσιονομικές πολιτικές είναι και οι ευκαιρίες η διαφάνεια και η σιγουριά που προσδίδουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε ένα κράτος που κάνει εκτεταμένη τη χρήση των νέων τεχνολογιών στις συναλλαγές του με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε αυτό. θα πρέπει αυτό να γίνει κατανοητό. έλλειμμα ηλεκτρονική διακυβέρνηση σημαίνει έλλειμμα ανταγωνισμού για τα κράτη μέλη και πέρα από την πρόβλεψη εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσα από τα διαρθρωτικά ταμεία θα πρέπει να υπάρξει και εκτεταμένη ανταλλαγή καλών βέλτιστων πρακτικών και εμπειριών στον τομέα αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ. E, και εγώ σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, η κυρία Μπασέσκου. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τη συνάδελφο Τσικόου για την θαυμάσια έκθεσή της. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες δίνουν ευκαιρίες για βελτίωση και εξυγχρονισμό των δημοσίων υπηρεσιών και των υπηρεσιών προς τον πολίτη και τις επιχειρήσεις. Αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια όσον αφορά τις διοικητικές δραστηριότητες. Ένα μεγάλο κομμάτι των δημοσίων υπηρεσιών ε, στα κράτη-μέλη αντιμετωπίζει προκλήσεις πλέον. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση μπορεί να οδηγήσει σε μεταρρύθμιση της δημόσιας υπηρεσίας ώστε να καταστεί θετικό συντελεστή της οικονομίας. Η οικονομία μπορεί να προχωρήσει με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Μπορούμε να ανταποκριθούμε καλύτερα στις προκλήσεις όλοι μας με αυτό. Πιστεύω ότι ο ευρωπαϊκός χώρος για διασυνοριακές συναλλαγές και για μικρομεσαίες θα βοηθήσει και την ενιαία αγορά. Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση βοηθάει και τους μη προνομιούχους. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μπάσκα. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα καταρχήν να χαιρετήσω τις προσπάθειες της εισηγητρίας, διότι προσπάθησε να ρίξει νέο φως σε αυτό το πρόβλημα ε, και ε, όσον αφορά την ε, ε, ε, τυποποίηση της πληροφορικής είναι πολύ σημαντικό τα συστήματα που χρησιμοποιούν οι πολίτες να επικοινωνούν μεταξύ τους διότι τώρα έχουμε τα συστήματα της Microsoft, Android και σε ορισμένα μηχανήματα δεν λειτουργούν σωστά γι' αυτό και θα πρέπει να έχουμε μία αρχή σε, ευρωπαϊκή, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο η οποία θα εξασφαλίσει την ε, ε, λειτουργία μεταξύ των συστημάτων αυτών. Ευχαριστώ. Κύριο Σαγκεντίνο, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα πρέπει όμως να μειώσουμε την γραφειοκρατία, να επιταχύνουμε ε, την πρόοδο και να κάνουμε και οικονομίες. Σχετικά με αυτά που είπε η κυρία Τίκαου ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν το 90% των επιχειρήσεων δείχνει ότι πρέπει να υπάρξει ψηφιακή τεχνολογία η οποία θα συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων διότι χρειάζεται μία ενιαία αντιμετώπιση αλλά η συγκεντρική Ευρώπη υπάρχει μεγάλη οπισθοδρόμηση δεν υπάρχει μία ενιαία αντιμετώπιση και θα πρέπει να προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα έχω ορισμένες επιφυλάξεις σχετικά με τους στόχους αυτούς καταρχήν θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων που είναι πολύ σημαντική για τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες και κατά δεύτερον λόγον θα πρέπει να υπάρχει μόνο αντιμετώπιση μέσα στη χώρα με αυτά τα στοιχεία. Ε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, η τεχνολογία επικοινωνίας ε, και πληροφόρησης που ανέφερε η συγγήτρια είναι ένα βασικό συστατικό της ε, σημερινής ζωής και επηρεάζουν και την οικονομική ζωή. 5% του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, οφείλεται στον τομέα αυτό της πληροφορικής που έχει ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες οι οποίες δεν έχουν ακόμη τύχη της σωστη εκμετάλλευσης διότι η ενιαία ψηφιακή αγορά δεν υπάρχει και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα ιδίως όσον αφορά την διασυνοριακή ε, παροχή υπηρεσιών στον ε, ψηφιακό χώρο και στον χώρο της πληροφορικής. Χρειάζονται αναπτύξεις και εξελίξεις στην ε, εσωτερική αγορά και επίλυση όλων των προβλημάτων. Ο κύριος Σόντι, επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τη συνάδελφο Τικάου για το πολύ σημαντικό έργο που πραγματοποίησε στην Επιτροπή Βιομηχανίας ε, για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ την Κομισιόν επίσης για το έργο της. Τρία σχόλια. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εξασφαλίσουμε την κάλυψη για τη δημιουργία όλων αυτών των τεχνολογιών σε ολόκληρη την Ήπειρο. Είναι αυτό στοιχείο ανταγωνίστικος. Στην Κορέζα, από την οποία ε, εκλέγομαι και στο Λιμουζάν δεν καλύπτονται από την τεχνολογία, από τους παρόχους όλα τα εδάφη και αυτό ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να έχουμε 100% κάλυψη. Δεύτερον, επειδή απλουστεύουμε τη ζωή, δεν πρέπει να γίνεται πιο περίπλοκη η δημόσια διοίκηση. Οι πολίτες έχουν κουραστεί από τη γραφειοκρατία. Και ένα σχόλιο όσον αφορά τους υπαλλήλους. Αυτές οι νέες τεχνολογίες πρέπει να μας δώσουν τη δυνατότητα να αφήσουμε τους υπαλλήλους τους εκεί που είναι και να μπορέσουν να συνδέονται με την κεντρική διοίκηση. Πρόεδρος, ο κύριος Κάλλη είναι ο επόμενος ομιλητής. Και θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Τίκα, που μας έδωσε μια πολύ σωστή σύνοψη ε, του πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Η αγορά η ηλεκτρονική έχει να κάνει με ανταγωνιστικότητα, με τον, τον ψηφιακό χαρακτήρα και αυτά είναι εξίσου σημαντικά. Βέβαια, εχμή του δώρατος λέμε ότι είναι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Σωστό είναι αυτό, και δίνει και τη δυνατότητα ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Δυστυχώς, 75% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν μπορούν να εμπορευτούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και ένα μεγάλο ποσοστό δεν εμπορεύεται έξω από τη χώρα τους. Όπως είπε ο Πιέρ Οντί, το πιο σημαντικό που πρέπει να κάνουμε είναι να έχουμε ευρυζωνική μεγάλη ταχύτητα διασύνδεση σε όλη την Ευρώπη και έτσι θα δημιουργήσουμε μια πραγματικά ενιαία αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ο τελευταίο ομιλητή είναι ο κ. Ματσαλά. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης ε, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι μια ευκαιρία να εξυγχρονιστεί το ε, σύστημα δημόσια διοίκηση στην Ευρώπη, μειώνοντα το κόστο, δημιουργώντα κίνητρα για την ανάπτυξη και τη γενοτομία σε επίπεδο περιφερειών. Η ηλεκτρονική τεχνολογία που χρησιμοποιείται στον τομέα της δημόσιας διοίκησης θα αυξήσει τη διαφάνεια, την ε, λογοδοσία και θα μειώσει το διοικητικό αυτό. Σε ορισμένε χώρε μέλη θα ταυτιστεί με την εξάλληψη εμποδίων στο δρόμο της διοικητική μεταρρύθμιση. Θα πλουστεύσει τι διαδικασίε σε διάφορα, σε διάφορα διοικητικά επίπεδα. Βεβαίω, χρειαζόμαστε μια σειρά από κανόνε για κρατικέ προμήθειε. Χρειαζόμαστε τυποποίηση και τη ρύθμιση νομικών θεμάτων που αφορούν την ηλεκτρονική υπογραφή και την άλλη ε, ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Βρέθηκα αντιμέτωπο με δυσκολίε όταν προσπάθησα να εφαρμόσω κάτι τέτοιο στη χώρα μου και για τον λόγο αυτό θα ήθελα επιμείνω ότι υπάρχει ανάγκη να βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε διαλειτουργικέ διακρατικέ υπηρεσίε. Όταν... Ε, θα ήθελα να συγχαρώ τον απειλητή για την εξαίρετη εισήγηση. Ευχαριστώ. Συμπερασματικά θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο. Δεν θέλω να ευχαριστήσω την κυρία Τίκο για την έκθεση για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Νομίζω ότι υποβάλλεται την κατάλληλη στιγμή και θέτει την ηλεκτρονική διακυβέρνηση στα πλαίσια ε, μια ψηφιακή, ενό ψηφιακού διαγράμματο. Βεβαίω συμφωνούμε ότι είναι μια ευκαιρία για να εξυγχρονίσουμε τον δημόσιο τομέα και να γίνει πιο φιλικό προ το χρήστη. Πολύ σωστά υπογραμμίσατε στην έκθεσή σας τη δύναμη που έχει ο τομέας του, της, ε, το ψηφιακό τομέα στην ε, Ευρώπη. Το συγκρίνεται με το, με το ΑΕΠ, με την ε, αξία στην αγορά και είπατε ότι συμβάλλει κατά 50% στην αύξηση της παραγωγικότητας. Φαντάζεστε λοιπόν το δυναμικό αυτής ψηφιακής αγοράς. Φαντάζεστε τι θα συμβεί αν εξαλειφθούν όλα τα προσκόμματα που υπάρχουν στις μέρες μας. Σε προσκόμματα που αντιμετωπίζουν και επιχειρηματίες και οι πολίτες όταν θέλουν να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες άλλης χώρας. Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο είπε σε επίπεδο ευρωπαϊκή συνεργασία θα καταβάλει προσπάθεια να ενισχύσει το πρόγραμμα δράση του 2015 και θα υποβάλει επανευρωπαϊκό πλαίσιο για την ηλεκτρονική ταυτοποίηση ελέγχου και ελέγχου, ελέγχου τη ιδιωσιότητα τη υπογραφή και τη υπογραφή. Καταρχά, θα πρέπει να μετεθεί το θέμα τη διαλειτουργικότητα και τη ορατότητα, αλλά και να εξαλειφθούν τα, εμπόρια, τα εμπόδια, αλλά και για να αντιμετωπιστούν ανάγκε που αφορούν την αμοιβαία αναγνώριση και και αποδοχή ηλεκτρονικής ε, ταυτοποίησης. Βεβαίως υποστηρίζουμε τις προσπάθειές σας ε, να γίνει πάγια τακτική ηλεκτρονική τιμολόγηση, τιμολόγηση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις ανάγκες των μικρομεσαίων ε, υπηρεσιών. Επίσης λαμβάνουμε υπόψη μας την φιλόδοξη έκκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, στις, στις ε, χώρες μέλη να καταστήσουν την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση. Αυτό που χρηματοδοτείται και δεν είναι ε, λιγότερο σημαντικό είναι η χρηματοδότηση σε ό,τι αφορά τι ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά δημόσια έργα, την ηλεκτρονική δημόσια γη, ηλεκτρονική ε, δικαιοσύνη. Για να μπορέσουμε να τα επιτύχουμε όλα αυτά ε, απαιτείται συνεργασία και βεβαίως ο στόχο είναι να επιτύχουμε μια ενιαία ψηφιακή αγορά η οποία θα είναι φιλική προ το χρήστη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Αυτό σήμανε και το τέλος της συζήτησής μας. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα αύριο.